πολιτική, το εμπόριο, τη δημιουργία ικανοτήτων ε, σε όλες τις περιοχές του κόσμου να ενισχύσουμε όλα αυτά τα σημεία και τις πτυχές αλλά να ενισχύσουμε ταυτόχρονα και τα εξωτερικά μας σύνορα και κυρίως το σύνορο Ελλάδας-Τουρκίας και αυτό είναι θέμα δημιουργεί προβλήματα στην Μεσόγειο και στα Δυτικά Βαλκάνια. Δεν θέλουμε η Κροατία να γίνει ένα άτυπο hot spot κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης. Θέλουμε δεν θέλουμε άλλες χώρες να ορθώσουν φραγμούς, ε, σειρματοπλέγματα, να κατασκευάσουν τείχους. Όχι. Με 6.500 αστυνομικούς προστατεύουμε τα σύνορά μας. Και προστατεύουμε τα σύνορα της Κροατίας και στο μέλλον τα, σύνορα του Σέγγιν και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θα πρέπει να εφαρμόσουμε το δίκαιό μας, ε, τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και τις διεθνείς συμβάσεις. Και οποιοδήποτε ισχυρισμοί για παραπτώματα θα διερευνηθούν και θα επιβληθούν κυρώσεις. Αλλά δεν θα πρέπει αυτοί οι ισχυρισμοί να θεωρούνται γενικευμένοι. Έχω επισκεφθεί τα σύνορα Κροατίας και Βοσνίας Αρεζεγοβίνης και όποιος άλλος τα έχει επισκεφτεί βλέπει πώς είναι τα πράγματα εκεί και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Frontex, να αλληλοβοηθηθούμε και να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το θέμα. Σε ό,τι αφορά τη διεύρυνση που ανέφερε ο κύριος Μπέι, θα ήθελα να πω το εξής δεν προσπαθούμε ε, να σπεύσουμε. Ε, για, απλώς εφαρμόζουμε μία ε, λογική υπεύθυνη για τις γειτονικέ μας χώρες. Γιατί οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν έχουν που να πάνε. Δεν πρόκειται να γίνουν ούτε μέλη των Ηνωμένων Πολιτειών, ούτε της Κίνας, ούτε α, της Ρωσίας ο μόνος, η μόνη τους διέξοδος είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να σφυριλατήσουμε και να διαρθρώσουμε σωστά τις σχέσεις μας και να τους δώσουμε την εντύπωση ότι θα μένουν ε, μονίμως ε, ε, στο προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χάσουν τη φόρο που έχουν πάρει για τις μεταρρυθμίσεις. Έναρξη διαπραγματεύσεων δεν σημαίνει κιόλα ένταξη. Θα χρειαστεί να εκπληρώσουν πολύ σοβαρούς όρους και προϋποθέσεις. Αλλά απλώς με την ένταξη διαπραγματεύσεων θα βοηθήσουμε αυτέ τι χώρε να επιταχύνουν τι μεταρρυθμίσει του. Και στη Σύνοδο Κορυφή του Ζάγκρεπ ελπίζω να έχουμε μια επιτυχή διακήρυξη που θα χαράζει το δρόμο για την επόμενη δεκαετία. Αυτό είναι ο στόχο μα. Κύριε σα ευχαριστώ για τι προτάσει σα και είμαι ευγνώμων που μα ε, ε, ευχηθήκατε καλή επιτυχία. Θα συνεργαστούμε μαζί σα για να την υλοποιήσουμε. Και όπω είπατε, δεν θέλουμε να είναι μια απλώ εορταστική ή τυπική προεδρία. Θα συνεχίσουμε το έργο μας. Έχουμε ήδη κάνει μια πολύ σοβαρή προεργασία και πολύ αφιερώνουν τεράστιο χρόνο ε, εργόδεις προσπάθειες για να προωθήσουν το ρόλο της Κροατίας και να ενισχύσουν τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι το προσεγγίζουμε. Ε, και για τη χρηματοδότηση, κύριε Κολακούσιτς. Διότι να, ισορροπία μεταξύ των παραδοσιακών πολιτικών μας και του εξυγχρονισμού. Δεν είναι μια απλή εξίσωση Ούτε κάτι εύκολο. Αν ήταν εύκολο, θα είχαμε ήδη επιτύχει συμφωνία για το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Ήδη από την προηγούμενη ίσω κοινοβουλευτική θητεία και την προηγούμενη επιτροπή φέρουμε τεράστια ευθύνη, γιατί υπάρχει μεγάλη διάσταση απόψεων, αλλά θα πρέπει όλοι να κάνουμε μικρέ υποχωρήσει, ώστε να βγούμε όλοι κερδισμένοι, και οι χώρε μα και οι πολίτε μα. Αυτή θα είναι και κατευθυντήρια γραμμή, ο μύτο τη Αριάδνη για μα για τι επερχόμενε διαπραγματεύσει. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, Αντρέη. Α ξεκινήσουμε τώρα τη συζήτηση. Πρώτο ο κύριο Ρέσλερ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Αξιότιμε πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αξιότιμε πρόεδρε τη κυβέρνηση, κύριε και κύριοι. Είναι λίγο φαϊνότερο ότι ιστορικά και πολιτισμικά η Κροατία ανήκει στην Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, σχετικά πρόσφατα, στη γενιά των γονιών μου, η ελευθερία, η δημοκρατία, αλλά και η πλήρη συμμετοχή στην ευρωπαϊκή οικογένεια ήταν μόνο απόμακρε και αβέβαιε επιθυμίε. Γι' αυτό και η Κροατική προεδρία στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί μία ακόμη συμβολική βαθμίδα στην ριζική μεταμόρφωση της Κροατίας. Από το δύσκολο αγώνα ε, για την ελευθερία και την ανεξαρτησία που ξεκίνησε πριν από τρεις δεκαετίες όταν γεννήθηκα εγώ, φτάσαμε στην ε, επιτυχή συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και σήμερα στην αρχή του νέου θεσμικού κύκλου έχουμε κοινού στόχου, αλλά ταυτόχρονα και κοινέ προκλήσεις που έχουν αναγνωριστεί και από τις προτεραιότητε τη Κροατική Προεδρία. Ένα από τα κέρια ζητήματα θα είναι σίγουρα η συμφωνία για το Πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Με τον εξυγχρονισμό της Ευρώπης δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να ξεχάσουμε τις παραδοσιακές και επιτυχημένες ε, πολιτικές, διαρθρωτικές πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης που στόχο έχουν τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και ανισορροπιών που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν. Πάντως είμαι πεπισμένος ότι η Κροατία με τη μοναδική της προοπτική θα συμβάλλει στη διευθέτηση και στην αντιμετώπιση των νέων και σημαντικών προκλήσεων στο επίπεδο της ασφάλειας, το τεχνολογικό, το κοινωνικό και το πολιτικό. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα είμαστε μια επιτυχής προεδρία για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να έχουμε μια ισχυρή Ευρώπη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσεις. Κυρία Μπόρσον, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η Κροατία αναλαμβάνει την, προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε δύσκολους καιρούς και παρά τις διαφορές μεταξύ μας, η ποιότητα ζωή των συμπολιτών μας θα πρέπει να είναι η προτεραιότητά μας. Στην κοινή ευρωπαϊκή αγορά κανένας δεν θα πρέπει να είναι πολίτης δεύτερης κατηγορίας. Η αγορά εργασία θα πρέπει να είναι ανοιχτή για όλους ε, όσοι θέλουν με τον καρπό της εργασίας τους να ζουν αξιοπρεπώς. Θα πρέπει να δώσουμε νέα όθηση στην εγγύηση για του νέου να διευκολύνουμε του επιχειρηματίες που θέλουν να επεκτείνουν τις ε, επιχειρήσεις τους και ε, διασυνοριακά και να εξασφαλίσουμε κατώτατο ευρωπαϊκό μισθό. Γιατί η εργασία κάθε πολίτη ε, έχει την ίδια αξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να αμείβεται ισότιμα. Δεν είμαστε άλλωστε μια κοινότητα ισοτήμων. Επίσης, όλα τα οικονομικά εργαλεία και μηχανισμοί θα πρέπει να έχουν μια μακροπρόθεσμη προοπτική και θα πρέπει να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία για να κοιτάξει πέρα από το κέρδος της και να αναλάβει την κοινωνική της ευθύνη. Επίσης, ε, να σκεφτούμε τους καταναλωτές που είναι η αδύναμη πλευρά στην αγορά. Θέλουμε υγιεινά και ποιοτικά τρόφιμα. Αυτό είναι προτεραιότητα, δεδομένου ότι έχουμε επιδημία παχυσαρκίας και πάχους με τις ε, αντίστοιχες ασθένειες που συνεπιφέρουν. Ε, χαίρομαι λοιπόν που δίνεται προτεραιότητα σε, πολιτικά, σε ποιοτικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ασφάλεια της διατροφής. Και θα πρέπει να γίνει το πρώτο βήμα για να έχουμε τα, τις σωστές διατάξεις που εδώ και να μήνα καθυστερούμε να τις εφαρμόσουμε στην Κροατία για τα ποιοτικά τρόφιμα. Σας εύχομαι καλή τύχη για την οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώπης χάρη των πολιτών μας. Για ένα λεπτό τώρα το λόγο έχει ο κύριο Φλέγκο. Σας ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε της ε, Κροατικής Κυβέρνησης, η άσκηση της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε τόσο δύσκολους καιρούς είναι για μια μικρή χώρα τεράστια πρόκληση. Και γι' αυτό θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή τύχη και καλή επιτυχία στην Προεδρία σας. Δεν θα ήθελα να ε, θυμηθούν την Κροατία ως ε, η η χώρα που άσκησε την Προεδρία όταν μια άλλη χώρα μέλος αποχώρησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ιδεώδης περίπτωση για νέες ιδέες, για νέα πρόοδο, για νέα βήματα. Και από αυτά που ακούσαμε σήμερα δεν άκουσα τον όρο παιδεία. Γιατί δεν δίνουμε έμφαση στην παιδεία. Και μετά τη διακήρυξη της Μπολόνια θέλουμε νέα πρόοδο, κυρίως τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Γι' αυτό προτείνω να διευρύνουμε τη διαδικασία της Μπολόνια ώστε να καλύπτει και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ώστε να έχουμε πιο ανταγωνιστική και πιο εναρμονισμένη γνώση και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δώσουμε περισσότερη έμφαση στην παιδεία και αυτό περιμένω από σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Κύριος το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, με μεγάλη χαρά σας ξαναβλέπω σε αυτό το νέο σας ρόλο. Και δύο θέματα θα ήθελα να σας θέσω. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε μία πρόταση για να υπάρχει διαφάνεια για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους απλούς πολίτες που πληρώνουν φόρους. Ε, ε, πραγματικά είναι πολύ άσχημο να βλέπουν τις μεγάλες εταιρείε να μην πληρώνουν φόρους. Θα το επαναφέρω το θέμα αυτό ε, στο θεματολόγιο του Ευρωπαϊκού Συμβούλου. Δεν προβλέπεται κάποια συνάντηση μέχρι στιγμής. Θα ήθελα λοιπόν να ξαναμπεί στην μερική διάταξη το θέμα αυτό να ολοκληρωθεί αυτό που ξεκίνησε η Φιλανδική Προεδρία και ελπίζω να υπάρξει πλειοψηφία σε επίπεδο Συμβουλίο. Επίση, όπω και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πλένκοβιτ, η Φιλανδική Προεδρία άρχισε να δημοσιεύει και τι τις συναντήσει ε, τη αντιπροσωπεία ε, στο πλαίσιο τη μη σύγκρουση συμφερόντων. Το κάνουν και άλλοι, η δική σα Προεδρία δεν το κάνει. Ακολουθήστε το φιλανδικό παράδειγμα, είναι μια πολύ καλή ιδέα. Ευχαριστώ. Η ε, κυρία Κόντε για 1,5 λεπτό. Desidero innanzitutto θα ήθελα καταρχάς να ευχηθώ καλή επιτυχία στις εργασίες των Κροατών γειτόνων μα, με του οποίου μοιραζόμαστε μια καταπληκτική θάλασσα, την Αδριατική, που μα δίνει πολλά και καλά ψάρια. Αλλά βλέπουμε ότι ε, η αλληλεία στην περιοχή αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο πολλών περιοριστικών μέτρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε ότι είχαμε σημαντικέ περικοπέ ήδη από το 2020, όσον αφορά για παράδειγμα το 10% των ημερών που μπορούν να περάσουν οι αλληλεί που ψαρεύουν μετράτα στην ε, περιοχή αυτή. Καταλαβαίνετε ότι οι αποφάσει αυτέ είναι αποφάσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία αντί να έρθει εδώ πέρα να μιλήσει για το ζήτημα αυτό και να συναποφασίσει τελικά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφάσισε να λάβει δράση μόνο στο πλαίσιο τη Γενική Επιτροπή για την Αλία στην Μεσόγειο. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν σύσσωμη να αντιταχθούμε στι προσπάθειε αυτέ που γίνονται για να αποδυναμωθεί ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνουν κοινέ προσπάθειε από την Κροατία, την Ιλιατία και τη Σλοβενία για την Αλία στην Ιδρυτική Θάλασσα. Ελπίζω ότι πραγματικά θα καταφέρουμε μέσω του εξαμήνου αυτού να συμβάλλουμε Βάλουμε θετικά προκειμένου να προωθήσουμε τομεί όπω η αλία για τον εξυγχρονισμό, για παράδειγμα, των ελευτικών σκαφών. Καθότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι παρούσα, θα ήθελα να ζητήσω και το ακόλουθο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προτίθεται πραγματικά να προωθήσει περισσότερο ή τελικά να αποσύρει το πολιετές σχέδιο όσον αφορά την αλία πελαγικών ειδών στην Ιδρατική θάλασσα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε μέσω των σωστών αποφάσεων να προωθήσουμε την οικονομική ευημερία για του Ευρωπαίου πολίτε. Είναι πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να προωθήσουμε και μηχανισμού περιφερειακή συνεργασία όπω πρωτοβουλία Interreg. Σα ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας πενθυμίζω απλώς ότι θα πρέπει να μιλάτε λίγο πιο αργά για να μπορούν να παρακολουθούν και οι διερμηνείς. Ο κύριος Τέρτσου τρέχει το λόγο για ένα λεπτό. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πλένκοβιτς, ε, ε, σας ε, εύχομαι κάθε επιτυχία και σε σας προσωπικά και στην Προεδρία και πραγματικά με συγκινεί προσωπικά το ότι λαμβάνετε την Προεδρία διότι όταν ως δημοσιογράφος στις αρχές δεκαετίας του 90 μέσα στα χαρακόμματα και στα κατεστραμμένα σπίτια πτώσια στο Καρλόβα της Λαβωνία στην Κράινα ούτε καν μπορούσα να ονειρευτώ ότι θα μπορούσατε και να λαμβάνετε Προεδρία ως Κροατία ακριβώ επειδή είναι τόσο ωραία η επανένωση των Ευρωπαίων από το Τάλι μέχρι το Κάντιθ, από το Ζάγκρεπ μέχρι το Άμστερνταμ, δεν θα πρέπει να αποτύχει αυτή η επανένωση και μπορεί να βοηθήσει η κρατική Προεδρία λέγοντα και προειδοποιώντα ε, ότι δεν θα πρέπει να γίνει όμοιρο η Ευρώπη μια ε, σοσιαλδημοκρατική ιδεολογία που ουσιαστικά αγνοεί, καταστρέφει έθνη. Δεν θέλουμε ένα υπερκράτο, γιατί αυτό θα ε, θέσει τέλο στη δημοκρατία. Δεν θα πρέπει να επιβάλλονται παράλογα ιδεολογικά σχέδια όπω είναι το ε, Πράσινο Σύμφωνο ή αυτή η τόσο ύποπτη διάσκεψη για το μέλλον τη Ευρώπη ουσιαστικά θέλει να προσανατολίσει και να κοροϊδέψει τα ευρωπαϊκά κράτη. Είναι κάτι που προβλέπεται που δεν το θέλουν σίγουρα όλοι οι πολίτε τη Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό. Η κυρία ε, Μπιέρκ. Ένα λεπτό, κυρία Μπιέρκ, ναι. Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Πρωθυπουργέ Πλέγκοβιτς, εδώ είμαι. Λέει η Προεδρία σας ότι θέλετε να εστιάσετε στο κράτος δικαίου ε, και στην ε, ανθρώπινη μεταχείριση, διαχείριση της μετανάστευσης. Εγώ διάβασα τις σχετικές αναφορές και επισκέφθηκα ε, το νότιο τμήμα της Κροατίας, βόρειο τμήμα της Βοσνίας και πραγματικά είδαμε 10.000 αποθήσεις και 25.000 το 2019 και Έχοντας διαβάσει όλες τις αναφορές και τη βιαιότητα ε, από την ε, κροατική αστυνομία, πρέπει να σας πω ότι ε, πραγματικά άκουσα και πάρα, είδα και έμαθα και πολύ χειρότερα από αυτά που είχα διαβάσει. Ε, πάρα πολύ μεγάλη βιαιότητα, ε, φρικτά πράγματα. Ε, σίγουρα πρέπει να υπάρξει αλληλεγγύη προς πρόσφυγες και όχι να είναι στόχος επιθέσεων. Το μήνυμα πρέπει να είναι σαφές. Δεν υπάρχει κανένα κράτος μέλος που θα πρέπει στα σύνορά του να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο. Είναι κάτι απαράδεκτο. Το είπαν και άλλοι συνάδελφοι. Το είπε ο Μάρτιν Σίρντεβαν συγκεκριμένα. Θα πρέπει να υπάρξει μηχανισμός παρακολούθηση. Ε, και ελέγχου και θα πρέπει να είμαστε σαφεί και κατηγορηματικοί. Δεν μπορεί να γίνεται μέλο τη ε, περιοχή Σέγγεν αν δεν πάψει αυτή η κατάστασή Μπλε κάρτα έχετε, λέει η στη τη δέχεστε από τον κύριο Σόκορ. Ε, τη δέχεστε. 30 δευτερόλεπτα παρακαλώ έχετε. Ευχαριστώ. Γιατί λέτε ανακρίβειες και αναλήθειες, κύριε συνάδελφε. δεν... Ε, νομίζω ότι αυτό είναι προσπάθεια συκοφαντικής δυσφήμισης Κροατίας ε, και τέτοιες δηλώσεις δεν ε, είναι αληθείς. Δεν ξέρω από ποιες πηγές έχετε τέτοιες ανακριβείς πληροφορίες. Νομίζω ότι από τη στιγμή που δεν έχετε εξακριβώσει την αλήθεια των πληροφοριών που σας αναφέρετε, καλύτερα να μην τις υποβάλλετε αυτές τις πληροφορίες. Στο συγγνώμη, είναι γελίο αυτό που λέτε. Έχω διαβάσει τις εκθέσεις αυτές. Πραγματικά είδα και εγώ μόνη μου ότι υπήρχαν για παράδειγμα 20 μετανάστες οι οποίοι επαναπροωθήθηκαν βία από την κροατική αστυνομία. Η ίδια είδα πραγματικά ποια είναι η βία της αστυνομίας που αντιμετωπίζεται απέναντι στους μετανάστες αυτούς που επαναπροωθούνται προς τη Βοσνία. Επομένως μη λέτε δεν ισχύουν όλα αυτά. Ανταυτού πείτε μας πραγματικά θα κάνετε την απαραίτητη έρευνα, θα φροντίσετε την υπάρχει μια ανεξάρτητη επιτροπή προκειμένου να μην καταπατώνται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ο κύριο Σίντσιτ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Καταρχήν να δούμε ε, τι γίνεται με την Κροατία τη στιγμή που αναλαμβάνει την Προεδρία. Διαφθορά και αναρχία. Αυτή είναι η κατάσταση στην Κροατία σήμερα. Πριν από δύο χρόνια, ως ε, Εθνικός Βουλευτής, ε, είχα στείλει προφορική ερώτηση. Ήθελα πληροφορίες τι γίνεται με, την, με το κτίριο της ε, κυβέρνησης. Ε, ποιος ε, χρηματοδοτήθηκε για να κατασκευαστεί αυτό το κτίριο. Ακόμη απάντηση δεν έλαβα. Επίσης, είναι δημόσιο στοιχείο αυτό. Είστε υποχρεωμένοι να απαντήσετε. Ακόμη και στο δικαστήριο έχω προσφύγει, αλλά ακόμη δεν έχω λάβει, απόφαση, ε, δεν έχω λάβει απάντηση. Λίγα μέτρα πιο πέρα από την Κροατική Βουλή έχουμε ένα νέο κτίριο. Ε, δεν έχω πληροφορίες για αυτά που, τα, που σας ρώτησε. Αυτά δεν είναι έργο Πρωθυπουργού, αλλά απλού απαταιώνα. Γιατί λοιπόν έχουμε αυθαίρετα κτίρια και γιατί ε, στους συμμέτερους σας αναθέτετε τέτοια κονδύλια 5 εκατομμυρίων ευρώ και παραπάνω. Κυρία Νίμπλε, να Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, ε, κυρία Πρόεδρε τη Κομισιόν, κύριε Πρόεδρε Εύοντα ε, του Συμβουλίου. Είμαστε στην απαρχή μιας νέας χρονιάς, μιας νέας δεκαετίας και μιας νέας προεδρίας. Ε, και πραγματικά είστε πολύ τυχεροί ε, που ε, είσαστε εσείς στο πιδάλιο της Ένωσης. Σίγουρα αυτό έρχεται με πάρα πολλές προσδοκίες και εσείς μας δώσατε ένα πολύ θετικό, φιλόδοξο πρόγραμμα δραστηριοτήτων σε ό,τι αφορά τις μεγάλες προκλήσεις, τα μεγάλα ζητήματα. Θα ήθελα να μιλήσω λίγο για τη μετανάστευση. Εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2015 και μετά προσπαθούμε να εξεύρουμε κοινέ λύσεις. Και πράγματι στην αρχή της χρονιάς ε, γίνονται διάφορες εκδηλώσεις, ε, ε, παραδείγματος και στην Βαβαρία, στη χώρα. Και γίνονται πραγματικά πάρα πολύ αισθητέ οι φωνές των πολιτών που ζητούν κάτι να γίνει. Πραγματικά πρέπει και εσείς να βοηθήσετε να γίνει αυτή η τομή σε ό,τι αφορά την πολιτική ασύλου. Μαζί να αναλάβουμε τις ευθύνες μας για την αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης που είναι το μεταναστευτικό. Χρειάζεται ένα συνδυασμό. Να έχουμε ασφαλή εξωτερικά σύνορα, να έχουμε ε, μια ε, συντεταγμένη μετανάστευση και προστασία των προσφύγων και μεταναστών. Ε, βλέπω και ακούω τι λένε οι συνάδελφοι και για το Σέγγεν και για την μετανάστευση. Σίγουρα είναι κρίσιμη η κατάσταση ε, αν ακούσουμε τους Έλληνες αδέλφους ε, για το τι επικρατεί στα ελληνικά νησιά για παράδειγμα και για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο για την ε, Πράσινη Συμφωνία ακούστηκαν πολλά πάντως το φλέγον, το πιο φλέγον παραμένει η μετανάστευση παρακαλώ εστιάστε λοιπόν σε λύσεις τις οποίες θα πρέπει να δεχθούν όλα τα κράτη-μέλη. Ευχαριστώ. Η κυρία Πύριχ, το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Αξιότιμη, αξιότιμη Προεδρεύοντα, κύριε Πρωθυπουργέ, χαίρομαι πάρα πολύ που σας ξαναβλέπω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η κρίση στη Λιβύη, καθώς επίσης και η κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, καταδεικνύουν ότι η περιοχή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Θα πρέπει να προωθήσουμε την πολυμέρεια και τη διπλωματία με σαφεί δεσμεύσει. Γι' αυτό το λόγο είμαστε υπέρ των δεσμεύσεων τη Κροατική Προεδρία για μια ισχυρή Ευρώπη σε ένα κόσμο που βρήθη προκλήσεων. Είναι πολύ σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει πιο ισχυρή θέση στο διεθνέ προσκήνιο. Και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει όμω να μπορεί πραγματικά να πραγματοποιεί τι δεσμεύσει δεσμεύσει και τι υποσχέσει τη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και απέναντι στα Δυτικά Βαλκάνια. Θα πρέπει όλη η διαδικασία να είναι αξιόπιστη και θα πρέπει να ξεκινήσουν με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία οι ενταξιακέ διαπραγματεύσει ήδη από το Μάρτιο, πριν δηλαδή τη συνοδοκορυφή του Ζάγκρεμπ. Επίση, η Ευρωπαϊκή Ένωση καμία περίπτωση θα είναι ισχυρή αν υπονομεύεται η δημοκρατία. Για παράδειγμα, στην Πολωνία και την Ουγγαρία θα πρέπει να έχουμε σημαντική στεναρή δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου πραγματικά να προασπιστούν εκεί πέρα τα δημοκρατικά συστήματα. Για όλα αυτά τα ζητήματα, η δική μου πολιτική ομάδα θα βρίσκεται στο πλευρό τη Προεδρία. Σα. Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφοι. Ήδη έχουν εγγραφεί 16 ομιλητέ διαδικασία Eye. Θα κλείσω τον κατάλογο στο σημείο αυτό και δεν νομίζω θα καταφέρουμε να δώσουμε το λόγο και στους 16 ομιλητές. Είναι πολύ σημαντικό να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης. Πιέζει πάρα πολύ ο χρόνος. Όταν αρχίζει λοιπόν και φωτίζει με κόκκινους χαρακτήρες ο χρόνος θα πρέπει να ολοκληρώνεται. Η κυρία Αγέ έχει το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι η πέμπτη Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με το ακαθόδε ζήτημα του μελλοντικού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελπίσουμε ότι θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Ο Σαρλ Μισελ έχει προσπαθήσει και θα προσπαθήσει να βρει μία λύση, αλλά καθοριστικός ήταν και ο ρόλος που θα δώσει ο ρόλο τη κρατική προεδρία, Όσο καθυστερούμε, είναι οι Ευρωπαίοι πολίτε και κυρίω οι γεωργοί, οι περιφέρειέ μα, οι επιστήμονε και ερευνητέ μα, οι οποίοι ζημιώνονται. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε την απαραίτητη χρηματοδότηση. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποια θα είναι η χρηματοδότηση των προγραμμάτων και οι δικαιούχοι τι μπορούν να κάνουν στα πλαίσια αυτή τη αβεβαιότητα και από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πώ μπορούμε να διαπραγματευτούμε χωρί να γνωρίζουμε ποια θα είναι τα μέσα τα οποία θα διαθέτουμε. Κύριε Πρωθυπουργέ, είναι κοινό το μέλλον και κοινέ οι προκλήσει. Η καταπολέμηση κλιματικής αλλαγής δεν πρόκειται να δοθεί μόνο στο Λουξεμβούργο. Καταλαβαίνετε ότι η μετανάστευση δεν είναι μόνο ελληνικό ζήτημα. Δεν θα ασχοληθεί μόνο η Εστονία με την ψηφιακή επανάσταση. Είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε όλοι με ζητήματα και όχι μόνο για παράδειγμα η Γαλλία και η Γερμανία. Νομίζω ότι θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει τους δικούς τη ίδιους πόρους προκειμένου να τα βγάλει πέρα σε όλα αυτά τα ζητήματα. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μάρκαρτ έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρωθυπουργέ, και εγώ θέλω να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία για το εξάμεινο της Προεδρίας σας. Πραγματικά αναφερθήκατε σε σημαντικές προτεραιότητες, ε, προτεραιότητες και για μια Ευρώπη που ενώνει, είπατε. Και πραγματικά είναι πολύ σημαντικό σε αυτό το πλαίσιο να λάβουμε υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ε, και οι ισχυρισμοί για κάποιου πολιτικού ότι άλλα λένε και άλλα κάνουν. Θα πρέπει λοιπόν ε, αυτό που λέμε να το κάνουμε και πράξη, ό,τι αφορά την Ευρώπη που ενώνει, που συνδέει σε ό,τι αφορά ε, την πολιτική του ασύλου. Σίγουρα το επόμενο εξάμεινο και πιο μετά θα ανταλλάξουμε διαφορετικές απόψεις μεταξύ μας. Πρέπει όμως να είμαστε ειλικρινεί ε, τουλάχιστον και πραγματικά ανησυχώ διότι ε, το βλέπω και το έχω δει και στην Κροατία με τα ίδια μου τα μάτια ότι έχουμε τόσες πολλές αποδείξεις για αποθήσεις στα σύνορα και βίαιη μεταχείριση από τη μία αλλά από την άλλη πλευρά δεν ακούω να λέτε ναι θα το ερευνήσουμε, αλλά λέτε όχι δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θέλουμε επίση μια Ευρώπη λέτε που να προστατεύει. Δεν θα πρέπει να προστατεύει και τα δικαιώματα, ε, να τα ε, σέβεται και στα σύνορά τη. Αυτό θέλω να φροντίσετε. Ευχαριστώ πολύ Κύριο Μπαρντέλα, μισή λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Βλέπουμε ότι η χριστιανοδημοκρατική κυβέρνηση της Κροατίας αναλαμβάνοντας την εκπεριτροπής Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή προωθεί συγκεκριμένα ζητήματα και από ό,τι φαίνεται πολλές φορές με τις πράξεις της και γενικότερα μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης επεμβαίνει τελικά στις εθνικές πολιτικές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως κάναν και προηγούμενες Προεδρίες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανταυτού βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο οι Ευρωπαίοι πολίτες στην Ιταλία στην Ισπανία, στη Γαλλία αντιδρούν και δεν το θέλουν αυτό. Βλέπουμε ότι όλο και περισσότερο υπάρχουν κάποιε ομοσπονδιακέ φεντεραλιστικέ δυνάμει που θέλουν μεγαλύτερη ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιο αργά, λέει κυρία Πρόεδρο και που στρέφονται κατά τη εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Το 2013 εντάχθηκε η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπήρχε τότε μια έντονη θεσμική κρίση και βλέπουμε ότι επλήγησαν συγκεκριμένες, συγκεκριμένοι τομείς, όπως για παράδειγμα την αυπηγία της Κροατίας, τα οποία έπρεπε να ευθυγραμμιστούν με τους κοινοτικούς κανόνες. Δεν μπορείτε λοιπόν να τα γνωρείτε όλα αυτά, κύριε Πρωθυπουργέ. Τίποτα το πανταστατικό δεν έχει το πρόγραμμά σας και σαφώ δεν πρόκειται να αλλάξει την ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Και α μην ξεχνάμε ότι ακόμα και ο πρόεδρο Μακρόν θα λυγίσει υπό την πίεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά την απόφαση που θα πρέπει να ληφθεί, για παράδειγμα, για την Αλβανία, ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα, ιδίω στο μεταναστευτικό τομέα που προέρχονται από τη χώρα αυτή. Και νομίζω ότι ε, όλο και περισσότερο θα βλέπουμε ότι θα υπάρχει μία αδράνεια από πλευρά θεσμικών οργάνων που θα λειτουργεί κατά των Ευρωπαίων πολιτών. Ο κύριο Γιουρίτσα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ε, σημαντικό καθήκον της Ευρωπαϊκής της Κρατικής Προεδρίας είναι να εξασφαλίσει διεκπαιρέωση των διαπραγματεύσεων για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο. Αυτό θα είναι και πιο σημαντική της ευθύνη. Επίσης θα πρέπει να καλύψουμε το χρηματοδοτικό κενό που θα έχουμε Μερικοί προτείνουν αύξηση των εθνικών εισφορών. Δεν νομίζω όμως ότι η πρόταση για αύξηση φορών ή για νέους ευρωπαϊκούς φόρους είναι καλή λύση. Θα πρέπει να κάνουμε καλύτερη διαχείριση των ε, υπαρχών των πόρων. Η Σλοβακία είναι καθαρή δικαιούχος ε, παραλήπτης ευρωπαϊκών κονδυλίων. Αλλά ίσως ε, η λύση δεν είναι μόνο η περικοπή των δαπανών, γιατί Μέχρι στιγμής είχαμε την ίδια ψελίδα κατανομής των ευρωπαϊκών κονδύλιων παρά την αναποτελεσματικότητα που διαπιστώσαμε μερικές φορές. Θα ήθελα λοιπόν το Συμβούλιο να καθορίσει καλύτερα τους στόχους των πολιτικών και να ε, αξιολογήσει πιο κριτικά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων. Παπαδημούλης. Κυρία Φόρντερ Λάιεν, ας λέμε αλήθειες εδώ μέσα. Στην κρίση της Λιβύης και στην κρίση μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα, είναι ουραγός. Είμαστε ένας οικονομικός γίγαντας, αλλά ένας πολιτικός νάνος. Και κύριε Πλένκοβιτς, αν θέλουμε μια πιο ισχυρή Ευρώπη και στη διεθνή σκηνή, που να παίζει έναν ρόλο συντελεστή ειρήνης με πολιτικές και διπλωματικές λύσεις, πρέπει πολλά πράγματα να αλλάξουν και η προεδρία σας δεν θα κριθεί από τα ωραία λόγια θα κριθεί από το αποτέλεσμα στο τέλος του εξαμήνου. θα μπορέσετε να συμβάλλετε έτσι ώστε να εγκριθεί ο νέος πολιετής προϋπολογισμός με βάση τις προτάσεις του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου έτσι ώστε να μην έχουμε περικοπές στα κονδύλια της συνοχής ή στα κονδύλια για την περιφερειακή ανάπτυξη την καινοτομία. θα συμβάλλετε στο να ξεκινήσουν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις για τη βόρεια μακεδονία και την αλβανία τον μάρτιο θα μπορέσετε να εγκρίνετε το φάκελο μεταρρύθμισης των πολιτικών ασύλου που έχει ετοιμάσει εδώ και δύο χρόνια το κοινοβούλιο και η κομισιόν και μπλοκάρει στο συμβούλιο. από αυτά θα κριθείτε. Σας ευχαριστούμε κύριο Σκοράου για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλημέρα σας κυρία Φόρντελάιν, καλώς επιστρέψατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κύριε Πλένκοβιτς. Ακούσαμε τις προτεραιότητές σας και τις δεσμεύσεις σας προκειμένου να προωθήσετε περισσότερο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα ευρωπαϊκά νησιά, κυρίω όσον αφορά την κλιματική μετάβαση. Είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στα νησιά αυτά κατά τη διάρκεια τη εξάμηνη προεδρία σα. Αναφερθήκατε επίση σε επενδύσει στην κοινοτομία, την ψηφιοποίηση, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν νέε δεξιότητε που ανταποκρίνονται σε νέα νέε θέσει απασχόληση. Σαφώ θα πρέπει όλα αυτά να αντιμετωπιστούν στα πλαίσια τη νέα αυτή ε, ευρωπαϊκή πράσινη ε, εποχή. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να καταφέρουμε να απαλλάξουμε από του δημοσιονομικού περιορισμού τι λεγόμενε οικολογικέ πράσινε επενδύσει. Το πιο σημαντικό να καταφέρουμε οι θεωρητικοί μας στόχοι να γίνουν πραγματικά μέτρα, τα οποία θα οδηγήσουν όντως σε βελτίωση τη ζωή των Ευρωπαίων πολιτών. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην πρώτη σας Προεδρία. Σας ευχαριστούμε για 1,5 λεπτό. Κύριο Ευχαριστώ πολύ αξιότιμη κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ε, κύριε ε, Πρωθυπουργέ της Κροατίας. Θα μιλήσω για τη διεύρυνση. Χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί το θέσατε σε ε, προτεραιότητα πρέπει να πείσετε, και αυτό είναι δύσκολο εγχείρημα, για την νέα προσέγγιση στα κράτη-μέλη και δεύτερον να, ε, την, ε, να επαναφέρετε την εμπιστοσύνη στις, ε, στους πολίτες των Δυτικών Βαλκανίων για το μαστείο και το καρότο και πώς χρησιμοποιούνται αυτά. Η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών στηρίζουν ε, την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, αγαπούν την ευρωπαϊκή ιδέα, παρά το γεγονός ότι ε, φέρθηκε στα κακιά πεθερά πρόσφατα Ευρωπαϊκή Ένωση. Με εσά ε, στις ηγετικέ θέσεις, κυρία Φοντελάιν, κύριε Πλένκοβιτς, ίσως αυτά αλλάξουν. Η Ουγγαρία, εμείς οι Ούγγροι θέλουμε μια σταθερή, ευμερούσα γειτονία και θέλουμε και τα Δυτικά Βαλκάνια, γιατί χωρί αυτά δεν θα είμαστε αρκετά ισχυροί ω Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανθέξουμε ε, τι πιέσει ε, τη παγκόσμια πολιτική. Άρα στα χέρια σας ε, πλέον ε, είναι το μέλλον και η κατάσταση αυτή, κύριε Πρόεδρε Βοντα του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ε, υπάρχει αίτημα ε, από τον κύριο Λουίς Καρικάνο, ε, μπλε κάρτα συγκεκριμένα. Τη δέχεστε, κύριε Ντέλη. Μισό λεπτό. Όχι, υπάρχει κάποια σύγχυση. Δεν έχει ζητηθεί ε, μπλε κάρτα. Άρα προχωρούμε στον επόμενο, τον κύριο Ερτούγκ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Καλώ ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για μια ακόμη φορά και καλή τύχη στην Προεδρία σα. Θα ξεκινήσω ε, με μία φράση ε, λόγω του ότι μιλήσατε για τη συνθεσιμότητα. Και ε, επειδή αυτό θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να σα πω ότι παραμένουν περιοχές στην Ένωση που δεν έχουν ή έχουν πολύ περιορισμένη ε, συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο. Και αυτό επηρεάζει δύο στις αγροτικές περιοχές και περιοχές ε, ε, που πλήττονται από την απερίμωση. Όμως θα πρέπει όλες οι περιοχές ε, να έχουν τις δέουσες ψηφιακές υποδομές. Το 5G δεν είναι απλά ένα συνθηματικό, είναι η βάση για πάρα πολλές εφαρμογές, για τις επιχειρήσεις, για την υγεία, τις μεταφορές, την ενέργεια. Και αυτή η εμβαλωματική κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ένωση δεν είναι αποδεκτή. Γι' αυτό κυρία Φοντερ Λάιεν, στρέφομαι σε εσάς τώρα, κάτι πρέπει να γίνει για να αποφύγουμε τέτοιου είδους ε, ε, εμβαλωματικά ε, συμβαλωτικέ εικόνες στον τομέα του 5G, αυτή τη τεχνολογίας. Και επίσης δεν πρέπει να έχουμε μια κούρσα προ τα κάτω στα κοινωνικά και εργασιακά Σα ευχαριστώ και ξανά καλή επιτυχία στην Κροατία. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κυρία Τσέχ. Ευχαριστώ. Αγαπητοί φίλοι Κροάτε, Πολύ συχνά ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Τώρα εσεί θα διαλέξετε και θα μα προτείνετε τον δρόμο που συλλογικά θα ακολουθήσουμε. Γιατί σε τόσο κρίσιμου καιρού η καθοδήγηση θα είναι πολύ σημαντική. Έχουμε αυξανόμενε ανισότητε, κλιματικέ αλλαγέ, Brexit και προβλήματα με κράτο δικαίου σε μερικέ χώρε. Όλα αυτά είναι θέματα με μακροπρόθεσμε συνέπειε για το σύνολο τη Ευρωπαϊκή μα οικογένεια. Γι' αυτό σα παροτρύνω να μην υποτιμήσετε τη σημασία των τραγουστών διαδικασιών κράτους δικαίου. Δεν αφορά μόνο την Ουγγαρία το ζήτημα, αλλά το σύνολο της κοινότητάς μας. Γιατί θα πρέπει να δείξουμε τον αυτοσεβασμό και να κάνουμε κάτι όταν ψηφούνται οι κανόνες και οι αρχές μας. Και επίση θα πρέπει να ανακτήσουμε τον αυτοσεβασμό μα, γιατί πολύ συχνά λείπει δυστυχώ αυτό το χαρακτηριστικό. Και ελπίζω να έχετε το κουράγιο και την ε, αυτοπεποίθηση να δράσετε ω πρωταγωνιστή του κράτου δικαίου και να προωθήσετε το άρθρο 7 που έχει κάπω κολλήσει στο παρελθόν. Θα πρέπει να δώσετε λοιπόν το καλό παράδειγμα και να αφήσετε μια παρακαταθήκη που θα μα ε, χρησιμεύσει και στο μέλλον. Ευχαριστώ. Κυρία Στρίκ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να καλωσορίσω τη, τον Κροάτη Πρωθυπουργό και την Κρατική Προεδρία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εύχομαι και καλή επιτυχία για, τους, για την υλοποίηση των στόχων. Ένα στόχο είναι η υλοποίηση του Συμφώνου για το Άσυλο με βάση την αρχή τη ελεγγύη και το δικαίωμα στο άσυλο. Η οθέτηση όμω τη νέα νομοθεσία ίσω είναι πολύ χρονοβόρα, ίσω κρατήσει χρόνια ολόκληρα. Ευτυχώ βέβαια έχουμε αρκετέ διατάξει που ισχύουν και αν εφαρμόζονται σωστά ήδη θα οδηγούσαν σε μια εναρμόνιση του συστήματος. Οπότε θα ήθελα να ρωτήσω τι θα κάνει η Κροατική Προεδρία για να προωθήσει τη συμμόρφωση με το τρέχον και εκτιμένο για το άσυλο σε όλα τα κράτη-μέλη. Και μια από τις βασικές παραβιάσεις ε, που λαμβάνουν χώρα είναι οι επαναπροωθήσεις, ε, οι αποθήσεις που φαίνεται ότι γίνονται σε πολλά εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ως εισηγήτρια του, τη συνέλευση του Συμβουλίου τη Ευρώπη, ασχολήθηκα με τα θέματα αυτά και μάλιστα επισκέφθηκα και τα κροατικά σύνορα με τη Βοσνία. Και πραγματικά ε, συγκλονίστηκα και σοκαρίστηκα από τις ε, πολύ τεκμηριωμένες ε, υποθέσεις για βία επαναπροώθηση, απόθεση και ουσιαστικά απόρριψη της πρόσβασης σε μια διαδικασία χορηγής ασύλου. Τι σκοπεύει να κάνει η Κροατία ώστε να τεθεί ένα τέρμα σε τέτοιες πρακτικές και να καταπολεμηθεί αντίστοιχη εφαρμογή τους και σε αλλα κρατημέλη. Δυστυχώ έχετε υπερβεί το χρόνο αγόρευσή σα και έτσι στερείτε από άλλου συναδέλφου να λάβουν το λόγο. Θα είμαι πολύ αυστηρή λοιπόν στην τήρηση του χρόνου αγόρευση από εδώ και πέρα. Για 1,5 λεπτό ο κύριο Νταρέ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και τον Πρωθυπουργό Πλέκοβιτσα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε πάρα πολλέ προκλήσει. Το σλόγγαν σα είναι μια ισχυρή Ευρώπη σε ένα κόσμο προκλήσεων. Έχετε λοιπόν μια καταπληκτική ευκαιρία αλλά και μια πρόκληση μπροστά σα προκειμένου να ανακτήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτε την εμπιστοσύνη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να πείσετε εσεί του Ευρωπαίου πολίτε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί όχι για τα μεγάλα συμφέροντα, αλλά για του ίδιου του πολίτε. Και ότι πραγματικά λαμβάνει υπόψη την τοπική πραγματικότητα, αυτή που έχουμε δηλαδή σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Μια μεγάλη πρόκληση είναι το Brexit, μια άλλη πρόκληση είναι το πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο, αλλά και η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερε υποδομέ και περισσότερη ασφάλεια και περισσότερη επιρροή στο διεθνέ προσκήνιο. Αλλά και τα άλλα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Υποστήριξη τη ανταγωνιστικότητα τη γεωργία, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, του τοπικού και περιφερειακού επίπεδου, του βιώσιμου τουρισμού, τη συνεργασία τη μακροπεριφερειακή. Είναι πολύ σημαντικό επίση να προωθήσουμε τους στόχους τους οποίους προωθείται όσον αφορά την κινητικότητα των φοιτητών, των ερευνητών, των σπουδαστών, καθώς επίσης και την προστασία της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς επίσης και των αθλημάτων. Διακόπτη, Πρόεδρος. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά, ζητάει Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κατάλαβα, σας ζητώ συγγνώμη. Εγώ προέρχομαι από την περιφέρεια του Βένετο, όπου αντιμετωπίσαμε πάρα πολλές προκλήσεις πρόσφατα και υπάρχει μια πάρα πολύ σημαντική ε, πολιτισμική συγγένεια μεταξύ της περιφέρειας μου και της Κροατίας. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία και σας υπόσχομαι ότι θα έχετε την αμέριστη υποστήριξή μου. Σας ευχαριστούμε κύριος το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα εξ ονόματος αντιπροσωπείας μου να επικεντρωθώ σε τρεις βασικές σας προτεραιότητες. Το ζήτημα του μελλοντικού προπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, το ζήτημα της ψηφιοποίησης, το ζήτημα της έρευνας και της ανάπτυξης. Ξέρετε ότι ο κόσμος και η τεχνολογία δεν μπορεί να μας περιμένει. Αναφερθήκατε κύριε Πρωθυπουργέ στο καθεστώ τη Δημοκρατία, στην προάσπιση του κράτους δικαίου. Αναφερθήκατε επίσης στην προάσπιση των εξωτερικών συνόρων. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πέρα από αυτό όμω θα πρέπει να ασχοληθούμε και με το Brexit. Θα πρέπει να διασφαλίσουμε και μετά το Brexit, μετά την αποχώρηση του Μανου Βασιλείου, τη συνεργασία με τη χώρα αυτή και όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Αντιμετωπίζουμε εδώ μια καινούργια κατάσταση βλέπουμε ότι υπάρχει μια νέα δυναμική διαδικασία την οποία θα πρέπει να προωθήσουμε περισσότερο προκειμένου οι χώρες αυτές να έχουν μια πραγματική ευρωπαϊκή προοπτική. κυρία Φίλιπς έχει το λόγο. κυρία Φόντερ Λάιν, σας είδα να φεύγετε σήμερα από το ξενοδοχείο σας με όλη αυτή την αυτοκινητοπομπή και τους σωματοφύλακές σας. Μήπως θα μπορούσατε κι εσείς να με συνοδεύσετε αύριο το πρωί. Καλώς ήρθατε κύριε Πρωθυπουργέ. Πραγματικά είναι εντυπωσιακά όλα αυτά που μας είπατε. Περισσότερα χρήματα για τις πιο ασθενείς οικονομίες, ανοιχτά σύνορα, πρόθεση της υποψηφιότητα τη Βόρεια Μακεδονία και τη Αλβανία. Για ποιο λόγο να θέλουμε να προωθήσουμε τι πολιτικέ αυτέ. Είναι παράλογε εντελώ και θέλετε επίση να βάλετε και την Κροατία στο αποτυχημένο ευρώ. Κατά αυτόν τον τρόπο θα εγκλωβίσετε τη χώρα σα στα πλαίσια της Ευρωζώνης και θα μπορέσει να απελευθερώσει μόνο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Το ευρώ αντιμετωπίζει μια χαμηλή χαμηλή οικονομική απόδοση και πολύ σημαντική ανεργία. Μην ενταχθείτε λοιπόν στην Ευρωζώνη. Οι πολίτε θέλουν περισσότερη ελευθερία και δεν θέλουν αυτή τη στιγμή να δεσμεύονται και να εγκλωβίζονται στις, στη βούληση κάποιων σημαντικών κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν πραγματικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δείξει ότι μπορεί να μεταρρυθμιστεί και ότι δεν θα καταργήσει τελικά του κανονισμού και τι οδηγίε τη, θα υπάρχουν και πολλέ άλλε χώρε οι οποίε θα αποχωρήσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μποζάλε Πόντ για μισή λεπτό. Καλώ ήρθε στο σπίτι σου, Άντρε. Και μάλιστα ε, πιο νεαρό πρωθυπουργό σε, σε, σε νεότερε χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολύ θετικό μήνυμα. Ε, Νομίζω ότι θα πρέπει να αποφύγουμε ότι ε, μειώνει την αξιοπιστία μας και ανοίγει ε, την, την πόρτα σε, σε πιο σκοτεινές δυνάμεις και συμφέροντα στα Δυτικά Βαλκάνια. Όταν κλείσουμε την πόρτα στα Βαλκάνια θα αρχίσει η διάλυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η απεικοδόμησή της. Και μιλήσατε για το διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Μετά την οδύνη του Brexit θα πρέπει ε, να δείξουμε με το δάχτυλο τους εχθρούς της Ευρώπης, τους εθνικιστές, τους αυτονομιστές και αυτούς που προσπαθούν να μας διχάσουν. Ο εθνικισμός είναι ο εχθρός της ειρήνης. Και να μην είναι αλήθεια, όπω είπε, Αντρέη, ότι θα πρέπει να προσπίσουμε το κράτο δικαίου με νύχια και με δόντια, με όλε τι δυνάμει μα. Θα πρέπει να σεβαστούμε την ανεξαρτησία των δικαστών και των δικαστηρίων. Θα πρέπει να σεβαστούμε τι δικαστικέ αποφάσει. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να δεχθεί τι δικαστικέ αποφάσει. Και αν θέλει να αναγνωρίσει ότι σέβεται το κράτο δικαίου, θα πρέπει να δεχτεί τα αιτήματα των δικαστών και δικαστήριων. Και ελπίζω ε, να είναι η τελευταία φορά που θα έχουμε Brexit, να είναι το τελευταίο διαζύγιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Brexit να είναι η τελευταία νίκη του εθνικισμού. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Πίτσουλα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Κύριε Πρωθυπουργέ, Πρώτα απ' όλα νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που σε αυτή την αίθουσα συζητούμε την πρώτη Κροατική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και χαίρομαι που δίνεται ιδιαίτερη προτεραιότητα ε, στα νησιά, που δείχνουν πως μπορεί να είναι προπομπή της ενεργειακής μετάβασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία χώρα λοιπόν, όπως η Κροατία, με χίλια και νησιά, πώς θα ενισχύσει αυτή τη διαδικασία Χαίρομαι για την ε, πρότασή σας για την ανανέωση της ε, πολιτικής ε, διεύρυνσης με την διοργάνωση της διάσκεψης κορυφής του Ζάγκρεπ με τις χώρες των Δυτικών, των Δυτικών Βαλκανίων. Θα είμαι συγγητής για το θέμα αυτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μετά την απόρριψη των έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για την Βόρεια Μακεδονία και Αλβανία, επανήλθε το θέμα αυτό στην στη συζήτηση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Η Κροατία είναι το νεότερο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει τις πιο πρόσφατες εμπειρίες από την ένταξη. Ε, είναι πολύ δύσκολο ιδιαίτερα όταν έχουμε το βέτο άλλων χωρών. Φαίνεται ότι η Γαλλία κάνει μια μεταστροφή. Έχετε μηνύματα από άλλες χώρες που εσθενίστηκαν τη γαλλική θέση για τα Δυτικά Βαλκάνια. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Κιουτσούκ. Ε, ευχαριστώ πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κύριε Πλένκοβιτ, να συγχαρώ την Κροατική Προεδρία για το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα, ιδίω όσον αφορά τα Δυτικά Βαλκάνια. Πολύ φιλόδοξη έναρξη αυτή τη νέα αυτή χρονιά και για την κυρία Φόντερ Λάιεν, η οποία στο Ζάγκρεπ είπε ότι θα πρέπει να δοθεί πράσινο φω για την έναρξη των ταξικών διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία. Α αντλήσουμε όμω κάποια διδάγματα από την περσινή χρονιά. Α μην υποσχόμαστε καταρχά πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τηρήσουμε. Δεύτερον, Σήμερα η παγκόσμια πραγματικότητα είναι τέτοια που δεν μας επιτρέπει να διατηρούμε πλέον ε, τα Δυτικά Βαλκάνια στην πίσω αυλή, στον προθάλαμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει αμεσότατα και επιτακτικά οι χώρες αυτές να ενταχθούν συντομότατα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να αναλάβουμε επίσης πρωτοβουλίες, προκειμένου να καταλήξουμε σε μια νέα μεθοδολογία για την προσχώρηση των κρατών αυτών και άλλων κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να συμβουλευτούμε τις χώρες αυτές βέβαια διαφορετικά δεν θα ευοδοθεί όλη η διαδικασία. Και αυτό που μόλις τώρα είπε ο κύριος Πίτσουλα, η συνδιάσκεψη για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό και οι υποψήφιες χώρες να μπορούν να συμμετέχουν στη συνδιάσκεψη αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ και πάλι συγχαρητήρια κύριε Πλένκοβιτ. Σας παρακαλώ πολύ να τηρείτε το χρόνο αγόρευσης. Υπερβήκατε αυτή τη στιγμή κατά 20 δευτερόλεπτα χρόνο αγόρευσης και αυτό είναι υπερβολικό. Ο κύριος Κράτορα έχει το λόγο. 1,5 λεπτό. Κύριε Πρωθυπουργέ, σήμερα πριν από περίπου 28 χρόνια η Κροατία αναγνωρίστης και ως ανεξάρτητο κράτος από τα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη και τώρα κάθεστε εδώ και είστε ο Προεδρεύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία. Διαβάζοντα το πρόγραμμά σας πρέπει να σας πω όμως ότι απογοητεύτηκα κάπως. Μιλάτε για την υποψήφια προς ένταξη χώρα την Τουρκία. Θέλετε να πάρει και το κοσυφοπαίδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, και δεν ξέρω ε, αν είχε στηρίξει ο κύριος Τούτσμαν ε, αυτή την πολιτική τι θα είχε γίνει και αν θα την υποστήριζε και ο λαός της χώρας σας ουσιαστικά πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτικές ε, οι οποίες ε, θα συμβαδίζουν με τις προσδοκίες των πολιτών και όχι θα τις ε, διαψεύδουν. Βλέπετε τι γίνεται με την απογοήτευση του κόσμου για την Ευρώπη. Νομίζω ότι πρέπει να δώσουμε καλύτερες απαντήσεις απέναντι στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη. Αυτό κάνει η Κομισιόν, αυτό κάνει το Κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο μεγαλύτερος οικονομικός χώρος με τις χαμηλότερες ε, επιδόσει στον τομέα της ανάπτυξης και θα δαπανίσουμε τρία δις για την κλιματική αλλαγή, κάτι που ίσως να μην είναι τόσο ε, μια μελλοντική, σε κάτι που δεν είναι μια μελλοντική τεχνολογία κατά κάποιους. Ε, και εγώ περίμενα περισσότερα από, τον, από την Κροατία και όχι να επανέρχεται το φάντασμα της δεκαετίας του 90 η μεγάλο εντατικές ε, ε, προτάσεις, το ξέρετε πολύ καλά και εσείς από το παρελθόν σας, δεν φέρνουν τίποτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τωσανόφσκι. Κύριε Πρωθυπουργέ, το πρόγραμμα προτεραιοτήτων της Ευρωπαϊκής ε, Προεδρίας περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο για επικοινωνία, μεταφορές, ενέργεια και μιλάτε για την εφαρμογή και την πρόθεση της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Προσοχή όμως ε, κατά την εφαρμογή των ε, τωρινών μας στόχων, γιατί είναι περίπλοκη και από τεχνική και από οικονομική άποψη. Πολύ φοβάμαι ότι μετά την θέσπιση κάποιων στόχων για τη βιομηχανία, αμέσως θα φροντίσουμε να τους αυξήσουμε. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε στην ενίσχυση του προγράμματος Ορίζον Ευρώπη, προηγουμένως. Και αν δεν θέλουμε να αυξήσουμε ε, δυσανάλογα το κόστος της ενεργειακής μετάβασης, αυτό το μείζον ζήτημα δεν μπορεί να διευθετηθεί πριν ε, να λάβουμε και νέα επιστημονικά πορίσματα. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Ελπίζω να καταφέρετε να αυξήσετε τη χρηματοδότηση για το ορίζον Ευρώπη. Καλή επιτυχία στην Προεδρία. Ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Σπουσδεμόν. κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ. Χαίρομαι ιδιαίτερα που καλωσορίζω την Κροατική Προεδρία στο Συμβούλιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται μια χώρα που πρόσφατα ανέκτησε την ανεξαρτησία τη και έδειξε ότι είναι επάξιο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ευχαριστώ τον κύριο Πλένκοβιτ που τάχθηκε υπέρ του διαλόγου μεταξύ Ισπανία και Καταλωνία. Η Καταλωνία είναι σήμερα ένα εσωτερικό ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι παρούσα στη διάρκεια της κρατικής προεδρίας. Θα πρέπει να βρεθεί λοιπόν μια πολιτική λύση μέσω διαλόγου και διαπραγμάτευσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναζητήσει κοινού δημοκρατικούς μηχανισμούς για την αυτοδιάθεση και σίγουρα η καταπίεση, η καταστολή δεν είναι αποδεκτή λύση. Είναι και η ώρα για τους Ευρωπαίους πολιτικούς να υψώσουν τη φωνή τους και να δείξουν στον κόσμο ότι υπάρχει ένας καλύτερος τρόπος για και το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση είναι ο καλύτερο και πιο δημοκρατικό τρόπο για να επιληθούν εδαφικές διαμάχε. όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παντού στον κόσμο. Σα ευχαριστώ. Έχουμε δύο ε, ερωτήσεις μέσω της διαδικασία μπλε κάρτας. Τις δέχεστε? Όχι, λέει ο κύριος Πουτσιτεμόν. Ευχαριστώ. Επομένω, ε, απορρίφθηκαν τα αιτήματα και στρεφόμαστε στον επόμενο μιλητή. Για 1,5 λεπτό το λόγο, ο κύριο Μούρεσαν. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ Πλένκοβιτς, καλώς ήλθατε για μια ακόμη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χαιρόμαστε πολύ που θα ηγηθεί για έξι μήνες τη Ένωση. η χώρα σας, που είναι ένα παράδειγμα, ένα μοντέλο για τα Δυτικά Βαλκάνια. Υπό την ηγεσία σας ε, έχετε πετύχει οικονομική ευημερία ε, και πληρείτε, πληρούνται και πληρούνται όλα τα κριτήρια ε, για ε, την ε, προσχωρησία στην ε, ολοκληρωθεί αυτή η καλή προσπάθεια θα πρέπει να ε, γίνουν αντίστοιχε προσπάθειε από τι άλλε χώρε των Δυτικών Βαλκανίων και επίση θα πρέπει η Ένωση να σεβαστεί τι υποσχέσει που έχει δώσει στι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων και να του πει με ισχυρή φωνή ότι είστε μέρο τη Ένωση Ευρώπη, ανήκετε ε, στην Ευρώπη και θα γίνετε μέλη τη Ένωση. Οποιαδήποτε μπορεί να είναι δική σα συμβολή θα είναι ιστορική σημασία. Και επίση ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πλέκο, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα έχετε τη δυνατότητα αυτό να το δείξετε και στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων που θα έχουμε για τον προπολογισμό τη Ένωση. Η φιλοσοφία του Κοινοβουλίου για τι διαπραγματεύσει αυτέ είναι η εξή. Θέλουμε να χρηματοδοτηθούν επαρκώ και οι νυν και οι νέε προτεραιότητε. Προτεραιότητες γιατί είναι σημαντικέ και δεν είναι κάτι παροχημένο και έχουμε αποφασίσει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα για τι προτεραιότητε. Κατά πολέμηση τη κλιματική αλλαγή προστασία περιβάλλοντο, προστασία εξωτερικών συνόρων. Σταθείτε στο πλευρό του Κοινοβουλίου, σα παρακαλώ, και ε, πείτε και στου συναδέλφου σα ότι απαιτείται νοπό χρήμα. Πείτε στου ε, συναδέλφου από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ε, συνοδεύσουν τι δηλώσει του με πράξει, δίνοντα τους απαραίτητους πόρους και βοηθώντας βέβαια και στην σωστή δαπάνη αυτών των κονδυλίων. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντάνιελσον, για ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. ευχαριστήσω όμω και τον Πρωθυπουργό Πλένκοβιτ, ο οποίο μα παρουσίασε τι προτεραιότητε τη Κροατική Προεδρία. Η στιγμή αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική γιατί καθορίζουμε την πορεία που θα ακολουθήσουμε για τα επόμενα χρόνια. Εξ ονόματο πολιτική μου ομάδα, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να οικοδομήσουμε έναν πιο ισχυρό οικονομικό κοινωνικό πυλώνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Α μην ξεχνάμε ότι είναι πολλέ χιλιάδε οι Ευρωπαίοι πολίτε οι οποίοι χάνουν τη ζωή τους μέσω εργατικών ατυχημάτων. 8.000 επίσης ασθενούν από καρκίνο, ακριβώς επειδή εκτίθενται σε καρκινογόνες ουσίες στο χώρο εργασίας τους. Το Δεκέμβριο μάλιστα το Συμβούλιο ενέκρινε μια νέα στρατηγική προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα εργατικά ατυχήματα και προκειμένου να έχουμε μηδέν καρκίνους στο χώρο εργασίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν θα πρέπει να ακολουθήσουμε την πολιτική αυτή και ελπίζω πραγματικά ότι η Κροατική Προεδρία θα θέσει το ζήτημα των εργατικών ατυχημάτων και εργατικών θανάτων πολύ ψηλά στο θεματολόγιο τη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρουμε να έχουμε μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την υγεία και την ασφάλεια στον χώρο εργασία. Για ένα λεπτό, κυρία Μπιτζότο. Σα ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κουραστήκαμε πλέον, κουραστήκαμε από τι κενέ αυτέ δηλώσει τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η κατάσταση είναι έκρηθμη στη Λιβύη και παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση κοιμάται.

Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνει δράση. Έχουμε τρομοκράτες οι οποίοι απειλούν την ασφάλειά μας και παρόλα αυτά δίνουμε δισεκατομμύρια ευρώ στον Ισλαμιστή δικτάτορα Ερντογάν. Όλα αυτά μοιάζουν σαν ευγαλμένα από μια ταινία επιστημονικής φανταστίας και παρόλα αυτά αποτελούν πραγματικότητα εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εξακολουθούμε και χειροκροτούμε τη Μέρκελ, τον Μακρόν και εσά κυρία Φόντε Λάιεν. Τι άλλο πρέπει να συμβεί, τι άλλο πρέπει να συμβεί, τι άλλο άλλο περιμένουμε προκειμένου πραγματικά να λάβουμε δράση. Περιμένετε να βυθιστεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, ξυπνήστε. Διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει τη μοίρα του Τιτανικού. Σας ευχαριστώ. Για ένα λεπτό κύριος Ρος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει σταδιακά να καταργήσει τα ορυκτά καύσιμα. Αυτό όμω ε, δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, αιωλική, ηλιακή κτλ. Θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στο ενεργειακό μας μείγμα και την πυρηνική ενέργεια. Και μάλιστα είδαμε άρθρα ότι είναι πολύ δαπανηρή και μη βιώσιμη πυρηνική ενέργεια. Αντίθετα όμως, ε, οι ανεμογεννήτριες θα δημιουργήσουν τεράστια απόβλητα για το μέλλον. Χρειαζόμαστε πυρηνική ενέργεια και μάλιστα η τιμή της κιλοβατόρας με την πυρηνική ενέργεια στη χώρα μου είναι η μισή από ό,τι στη Γερμανία. Και, έχουμε, και η Γερμανία έχει παιδίσει 200 εκατομμύρια σε ΑΠΕ. τα αιωλικά πάρκα όμως και τα φωτοβολταϊκά δεν μπορούν να αντισταθμίσουν την σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων θα είναι πολύ δαπανηρή και χρονοβόρα διαδικασία. Θα πρέπει να είμαστε υπεύθυνοι σε επενδύσει. Και θα πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί και απέναντι στην Κίνα και τι Ηνωμένε Πολιτείε. Γιατί θα χάσουμε θέσει εργασία. Απευθύνω έκκληση λοιπόν στην κρατική προεδρία να, να επαναφέρει την πυρηνική ενέργεια στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόρμαν, ένα λεπτό, αξιότιμη πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιότιμη πρωθυπουργέ, ε, πραγματικά σας συγχαίρω για το πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα της πρώτης κρατικής προεδρίας και θα ήθελα να σας πω ότι είναι σημαντικό και σε ό,τι αφορά την ε, αγροτική ε, πολιτική, την πολιτική για την αγροτική ανάπτυξη, να την χρηματοδοτήσουμε επαρκώς μέσω του ΠΔΠ. Υπάρχουν αρκετές εκτάσεις και θα πρέπει λοιπόν να βοηθήσουμε τους αγρότες που κατοικούν και εργάζονται ε, σε αυτές τις περιοχές. Ε, δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε ότι και οι ε, αγρότες μας χρειάζονται την εισοδηματική στήριξη και μόνο αν είναι σε καλή κατάσταση θα παραμείνουν και εκεί οι αγρότες να εργαστούν και να ζήσουν και επίσης θα προσελκυστούν και νέοι. Θέλουμε λοιπόν επίσης να μην υπάρχει προσέλκυση ε, μόνο ε, πολύ μεγάλων επενδυτών, αλλά να υποστηριχθούν και οι ε, μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Ελπίζω με το πι και με τις αποφάσεις για την κοινή γεωργική πολιτική να μπορέσετε να διαμορφώσετε το μέλλον της Ευρωπαϊκής Γεωργίας προς το καλύτερο. Ευχαριστώ πολύ, Γιουγκέριους. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θέλω να συγχαρώ τον Πρωθυπουργό. Συγχαρητήρια γιατί πλέον έχετε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πρώτη φορά μετά την ένταξή σας. Βέβαια έχουμε στον ορίζοντα τον, τον Brexit και δεν πρέπει να λησμονούμε πως ο λόγος που έγινε Brexit ήταν που οι απλοί άνθρωποι ένιωθαν ότι δεν έχουν υποστήριξη Πρέπει λοιπόν από εδώ και πέρα να είμαστε φιλόδοξοι. Γι' αυτό θέλουμε και ένα φιλόδοξο και κοινωνικά υπεύθυνο πιδελταπή. Δυστυχώ δεν πάνε και τόσο καλά οι διαπραγματεύσει και είναι πολύ θετικό που ε, έχετε προτεραιότητα το ΠΔΠ. Θα πρέπει να πρικοδοτηθεί επαρκώ ο κοινωνικό πυλώνα. Πώ θα εξασφαλίσετε επαρκή χρηματοδότηση για την υλοποίηση του κοινωνικού πυλώνα. Γνωρίζω ότι είστε υπέρ της κοινωνικής αηφορίας. Δεν θα πρέπει να μείνει κανείς πίσω όμως. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για την κοινωνική πρόοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για ένα λεπτό κύριο Ρανζέλ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρωθυπουργέ, κυρία Πρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Καταρχάς θα ήθελα να χαιρετήσω την Κροατική Προεδρία και όλος ιδιαίτερος τον Πρωθυπουργό Πλένκοβιτς. Όχι μόνο γιατί η Κροατία είναι από τα νεότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί, αλλά γιατί ο Πρωθυπουργό Πλένκοβιτς είναι από τους πιο στρατευμένους ε, πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ του Ευρωπαϊκού Σχεδίου, είναι από τους πιο διάπειρους υπέρμαχους του Ευρωπαϊκού Σχεδίου και σας εύχομαι καλή επιτυχία στην Προεδρία και χαίρομαι για το άνοιγμα που κάνετε προ τα Δυτικά Βαλκάνια και χαίρομαι που στηρίζετε τι μεταρρυθμίσει των βαλκανικών χωρών που θέλουν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι που είναι σίγουρο είναι ότι δεν θα έχουμε Ευρώπη ή δεν υπάρχει Ευρώπη χωρί ένταξη και των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων στου κόλπους τη. Θα ήθελα επίση να χαιρετήσω την προτεραιότητα που δίνεται στη συνοχή και στο πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο. Και χαίρομαι για τις προσπάθειές σας υπέρ της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Γιατί υπήρχε αναφιβολία σαν το Συμβούλιο θα ε, προχωρούσε στην έναρξη της ε, διάσκεψης αυτής. Και χαίρομαι που η Κροατική Προεδρία θα στηρίξει στεναρά τη διοργάνωση της διάσκεψης για το μέλλον της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ζωχίνιο για ένα λεπτό. Μία ισχυρή Ευρώπη σε ένα κόσμο γεμάτο προκλήσει. Αυτό είναι το σύνθημα τη Κροατία για την πρώτη τη, την παρθενική τη Προεδρία στην, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σα εύχομαι καλή επιτυχία. Μία ισχυρή Ευρώπη όμω θα πρέπει να είναι μια Ευρώπη που θα έχει ικανότητα δράση και προόδου. Μία Ευρώπη ανάπτυξη θα πρέπει να έχει ένα φιλόδοξο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο χρηματοδότησης για να προωθήσει τη σύγκληση, τη συνοχή και να ενισχύσει τους ίδιους πόρους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μία ένωση που συνδέει θα πρέπει να, να προσετεριστεί τους πολίτες στο ε, μεγάλο σχέδιο δημοκρατίας και ειρήνης που αποτελεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με απαραίτητα μέσα για να το εφαρμόσει. Μία Ευρώπη που προτείνει θα πρέπει να έχει τη δικαιοσύνη ως σημείο αναφοράς και να, να αφήνει κανένα πίσω στους δύσκολους καιρούς. Και μία Ευρώπη με ισχυρή επιτροπή θα πρέπει να διατρανώνει τη θέση της ε, όχι μόνο μεταξύ ε, ισοτήμων που έχουν κοινέ αξίες αλλά κάνοντας συγκεκριμένα